Κύριε Βίλαντ. I have you, I have you for an explanation of... Έχετε δηλώσει ότι θέλετε να κάνετε μια επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Λένε. Καλώς, προχωρούμε. Ο κ. Σόσπακιουίτς έχει το λόγο. You have to push the button, Mr. Usbekic. You have to push the button. Για να μιλήσετε κύριε Ούσπαχιτ, πρέπει να πατήσετε πρώτα το κουμπάκι. Ε, ε, Πρόεδρε. Θέλω να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι υποστηρίζω αυτή την απόφαση. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω. Και τώρα επί της ουσίας, αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου της Επιτροπής για τις μικρομονάδες ή μικροεπιχειρήσεις και την υποχρέωση κατάθεσης ετησίων, ε, ετήσιων λογαριασμών. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται, που διεξάγεται σε διάφορα επίπεδα εξετάζεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις ε, κρατικές ε, εθνικές αρχές. Πρέπει να ισχύσουν κοινοί κανόνες, νομίζω, κοινοτικοί για όλους. Πρέπει ωστόσο να προβλέψουμε κάποιες ειδικέ διευκολύνσεις για τις μικρομονάδες χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και χωρίς να διαταραχθούν οι κανόνες του ανταγωνισμού. Ένας κοινό φόρος πρέπει να προβλεφθεί για τις μικρομονάδες ο οποίος θα μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη είτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις ή με βάση ε, άλλα κριτήρια. Συνάδελφοι, να σας πω κάτι. Οι επεξηγήσεις ψήφου είναι ένα λεπτό και εγώ και πεινάω κιόλα. Μην ξεπερνάτε την ώρα σα. Ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με την δυνατότητα η δυνατότητα απελευθέρωση των μονάδων από τους ετήσιους λογαριασμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μίλησε υπέρ της μείωσης της γραφειοκρατίας. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι είμαι υπέρ της ανάπτυξης ε, της ευρωπαϊκής ε, μεσαίας τάξης επειδή τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ε, μόνα τους για την απαλλαγή από την υποβολή ισολογισμού. Θεωρώ ότι πολλά κράτη συμπεριλαμβανομένης και τη Γερμανία, θα κάνουν χρήση αυτού του κανισμού. Έτσι λοιπόν με τον κανισμό αυτό δεν θα εξοικονομηθούν μόνο περίπου 2.000 ευρώ ανά επιχείρηση αλλά είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα για το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι είναι πολύ πιο φιλική προς τον πολίτη από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο ε, αυτού του παραδείγματος να ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Ο κύριος Μότι, ένα λεπτό. E Συνάδελφοι, δεν υποστήριξα την έκθεση, λένε ε, παρότι ασχολείται με μικρο που αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρώ ότι το ψήφισμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ε, για, λόγω των διαφορών ανταγωνιστικότητα μεταξύ επιχειρήσεων των κρατών μελών και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε, ιδίω σε μια εποχή κρίσεω. Κατόπιν η λειτουργία των λογαριασμών είναι ένα αναγκαστικό εργαλείο σημαντικό για να μετρήσει μια επιχείρηση στην αγορά και για να λάβει πίστοση από τι τράπεζε διότι με βάση τους λογαριασμούς ε, προσμετράται η καλή πορεία της διαχείρισης και των μικρών επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε περισσότερο με την ε, παροχή κινήτων στις μικροεπιχειρήσεις για να έχουν με μείωση φορολογίες που θα επιτρέπει στους νέους επιχειρηματίες να είναι πραγματικά ανταγωνιστικοί στην αγορά και θα τους επιτρέπει να παίρνουν ε, πιστώσεις από τα πιστοτικά ιδρύματα και να μην αυξάνονται οι ρυθμοί των ε, ανέργων. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή να υποστηρίξω την έκθεση Λένε που θα μειώσει το, το βάρος των διοικητικών διαδικασιών για τι μικροεπιχειρήσει. Θα μιλάμε για τι μικροεπιχειρήσει. Τονίζουν τη γραφειοκρατία που, και το γεγονό ότι πνίγονται κάτω από στίβε χαρτιών. Είναι λοιπόν λογικό οι μικροεπιχειρήσει να μην υπόκεινουν στου ίδιου κανόνε και κανονισμού όπω οι μεγαλύτερε επιχειρήσει. Νομίζω λοιπόν ήταν μια πολύ σωστή και υπεύθυνη απάντηση που δώσαμε σήμερα στις ανησυχίες των μικρών μονάδων στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή τροποποίησαμε ε, ε, μια νομοθεσία η οποία θα δημιουργήσει ένα καταλληλότερο επαγγελματικό περιβάλλον και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Θεωρώ λοιπόν το μια πολύ σωστή απόφαση. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο λένε όπως και άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο από κοντά και αυτό φάνηκε και σήμερα. Επίσης η πολιτική μας ομάδα ανέκαθεν θα στηρίξει τις ΜΜΕ, θεωρεί ότι είναι μια προτεραιότητα. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό το ότι το θέμα προωθήθηκε σήμερα και θέλουμε η γραφειοκρατία να μειωθεί αλλά και σχετικές δαπάνες για τις μικρομονάδες. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη βοήθεια για τις μικρές επιχειρήσεις. Τελειώνω για το πόσο ευέλικτη είναι η διάταξη αυτή, η οποία προσφέρει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ενσωματώσουν την οδηγία κατά την πλέον σκόπιμη στιγμή. Αυτό για να αποφευθεί οποιαδήποτε μορφή ε, παρανομίας που μπορεί να προκύψει από την ε, απρόβλεπτη μείωση του αριθμού των ελέγχων. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Το επόμενο. Πρόκειται για την Ευρώπη στον του 2020 και ο πρώτος ομιλητής είναι ο Φιλίπ Λαμπέρ για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο κύριε. Α, ε, η κυρία Λαμπέρ. Ο κύριος Λαμπέρ. Συνάδελφε κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η ψηφοφορία είναι κάτι το αξιοσημείωτο για δύο λόγου. Πρώτα πρώτα, οι τρει μεγάλε ομάδε αποφάσισαν να κάνουν αυτό το κοινό ψήφισμα και το κατέθεσαν έξι λεπτά πριν τη λήξη τη προθεσμία. Οπότε και ήταν αδύνατον εμεί να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τροπολογίε. Αυτό είναι παράδειγμα για το Κοινοβούλιο. Δεύτερη παρατήρηση. Μακάρι τελικά να έχει ένα νόημα αυτό το κείμενο με αυτή τη διαδικασία η Κομισιόν από τις ίδιες πολιτικές οικογένειες έχει ε, ε, πολιτικές στόχους και εμείς βγάζουμε αυτό το ψήφισμα που δεν λέει τίποτα πάνω στο τίποτα που δεν έχει πει η Κομισιόν και αυτό με την σύμπνοια των τριών μεγάλων οικογενειών αυτό βρεζιλεύει το Κοινοβούλιο ε, μας, μας, τίποτα δεν κάνουμε, λέμε το, το, το, το, το αυτονόητο. Ο επόμενος λέει ο πρόεδρος, Μανέσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτε θέλουν να υπάρχει πιο συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά την οικονομική πολιτική εν ώψη του 2020. Οπότε και εγώ θέλω να χαιρετήσω αυτή την αλλαγή πορείας που γίνεται όσον αφορά την οικονομική μας πολιτική και στρατηγική. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κάποιες πτυχές του θέματος δεν ε, εθίγησαν όσο και όπως θα έπρεπε. Οπότε σας επισημαίνω την προσοχή ότι όσον αφορά τη στρατηγία του 2020 δεν προκύπτει ακριβώς ποια είναι η σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και ε, στρατηγικής οικονομικής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε το πόσο σημαντική είναι η περιφέρεια, ο ρόλος περιφέρειας και να προσέξουν περιφερειακή πολιτική. Άρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συστρατευτούν, να προσέξουν την ε, στατηγική αυτή και να προσδώσουν τη σημασία που πρέπει εις τις τοπικές αρχές. Και τελικά η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από το πώς θα εμπλέξουμε τις ε, τοπικές αρχές σε εθνικό επίπεδο. Επόμενος, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ή στα πλαίσια του ατύπου Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου εγκρίθηκε αυτό το κείμενο με το οποίο θα βοηθηθούν οι αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προβλήματα τι σημαίνει όμως Ευρώπη ενώπιση του 2020, τι γίνεται με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρόκειται εδώ για μια απόφαση αλληλεγγύης. Και με την προοπτική του 2020 θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, να το δούμε πιο συγκεκριμένα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε την κάθε περιφέρεια με τις διορυθμίες της, τις της και θα πρέπει να δούμε το ότι θα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις με ταυτόχρονη σημασία πρέπει να προσδώσουμε στην ε, παιδεία και την έρευνα. Άρα να κάτσουμε και να δούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα κάθε περιφέρειας και κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για την προοπτική 2020. Επενδύσεις, παιδεία, διπλάσια πρικοδότηση πρέπει να δώσουμε και να προδούμε με τι υποδομές θα έχουμε καλύτερη γνώση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ο Παπα-Νικολάου για ενα Από, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε στο Κοινοβούλιο μας στις Βρυξέλλες καθώς και από τις τοποθετήσεις του Αρμοδίου Επιτρόπου και των αρχηγών των κρατών μελών αρκετών από αυτών στη συνέχεια προκύπτει ότι σε περιόδους κρίσης και όταν κάποια κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι απαραίτητη και στο πλαίσιο της νομισματική ένωση την οποία έχουμε είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη η χάραξη πολιτικών που θα διασφαλίζουν την αντιμετώπιση κερδοσκοπικών επιθέσεων κατά κάποιων συγκεκριμένων κρατών μελών. ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικέ οι τοποθετήσει που γίνονται αυτή την περίοδο σε σχέση με τη δημιουργία θεσμών και δομών ευρωπαϊκών για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων όπω για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. αναμένουμε πολλά από το συμβούλιο στη συνέχεια και με αυτή την προσδοκία ε, νομίζουμε ότι τα προβλήματα αυτή την κρίσιμη περίοδο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική μέχρι το 2020. Επί της αρχής οποιαδήποτε πρωτοβουλία για να βελτιώσει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηριχθεί. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να ασκούμε και κριτική. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική μέχρι το 2020 Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν πλέον όρια μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων. Δεν μιλάω βέβαια για ζητήματα όπως ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, η κληρονομιά. Αλλά όσον αφορά τα οικονομικά, η ευρωπαϊκή αγορά είναι μια κοινή αγορά. Εάν ίσχυε το αντίθετο, Αυτό θα σήμαινε πως ε, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στην ε, Ευρώπη θα είχαν διαφορετικούς κανόνες. Νομίζω λοιπόν ε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει κοινούς οικονομικούς όρους. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και των τεχνολογιών αλλά και να σημειώσουμε και την σημασία της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας έκοψα το μικρόφωνο. Η κυρία Γιάλα Σέντερ δεν φαίνεται πως είναι εδώ. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο για ένα λεπτό. Το κύριε Πρόεδρε. Η στρατη... Καταψήφισα την έκθεση γιατί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 βαδίζει στον ίδιο αποτυχημένο νεοφιλελεύθερο δρόμο της στρατηγικής της Λισαβόνας που οδήγησε στη διεύρυνση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στην αύξηση τη φτώχεια και τη ανεργία και αποτέλεσε βασική αιτία για την κρίση στην ευρωπαϊκή ένωση. επομένω απαιτείται ριζική αλλαγή του πλαισίου άσκηση οικονομική και κοινωνική πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο την πλήρη εργασία και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων. οι ηγέτε τη ευρωπαϊκή ένωση κατά το άτυπο συμβούλιο όταν ξέσπασε η κρίση κρύφτηκαν αφήνοντα κάθε κράτο να αντιμετωπίσει μόνο τα προβλήματα και τώρα έρχονται να επιτηρήσουν τα δημόσια οικονομικά ελλείμματα αντιμετώπισαν την ελλάδα ω το μαύρο πρόβατο και επιδιώκουν τη λήψη σκληρών μέτρων που θα λαμβάνονται σε βάρος των εργαζομένων της ελλάδας και των άλλων χωρών. επομένως απαιτείται η αντικατάσταση του αντικοινωνικού και αντιαναπτυξιακού συμφώνου σταθερότητα με ένα σύμφωνο ανάπτυξης και μεγέθυνση όπω το περιγράφει το ψήφισμα που κατέθεσε η ευρωπαϊκή αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα στρατηγική για να αντιδράσει στην οικονομική κρίση και σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής πρέπει να είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα όλων των ανθρώπων, φοιτητών, επιστημόνων, συνταξιούχων, πράγμα το οποίο αναφέρεται στο ψήφισμα Επίσης πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλιώς δεν θα βγούμε από την ε, κρίση. Κάποιοι θεωρούν πως δεν τονίζουμε αρκετά την πολιτική συνοχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί η έμφαση υπάρχει. Λέμε πως είναι σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης. Εάν όμως δεν εφαρμοστεί, καμία στρατηγική δεν θα μας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ, κύριος Μονσινιόρε. Καλημέρα κύριε Μονσινιόρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στιγμή να γίνει, είναι η στιγμή να δικαιωθούμε πολιτικά. Η κρίση έδειξε την αναγκαιότητα που υπάρχει να έχουμε περισσότερο συντονισμό. Θα πρέπει να αποκτήσουμε κύρωση οι διάφοροι φορεί, περισσότεροι φορεί, πόροι να δοθούν για τις υποδομέ, πραγματική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα πρέπει ε, να προχωρηθεί η ενοποίηση τη εσωτερική αγορά και θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή οικονομική φορολογική πολιτική. Κάποιοι έκαναν να μην βλέπουν τα διάφορα προϊόντα που πουλούσαν οι Αμερικανικές τράπεζες και δημιουργήθηκαν παρόμοια προβλήματα εντός Ευρωπαϊκής Ενώσης. Είναι ώρα τη ευθύνη και του θάρρου. Το ψήφισμα που ψήφισα με την ομάδα μου εμπεριέχει κάποια τέτοια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι ο Μπαρόσο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν περισσότερο θάρρο Ευχαριστώ. Και τέλος, ο κύριος Τσανέσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αυτή η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 είναι νεότερο αδελφάκι της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Αν δεν μαθαίνει κανείς από τον πιο μεγάλο του αδελφό δεν περνάει τις εξετάσεις και θα μπορεί να μελετήσει αργότερα. Ταυτόχρονα, όταν οι ηγέτες της Ευρώπης συζητούσαν την ανάγκη έγκρισης της στρατηγικής της τα κράτη-μέλη μείωναν τις δυνατότητες ελεύθερης διακίνησης ατόμων εργαζομένων και υπηρεσιών. Αυτή η νέα στρατηγική είναι κάπως καλύτερη από την εκδοχή που είχαμε πριν από δύο μήνες, όταν δεν αναφερόμασταν καθόλου στην συνοχή. Παρόλα αυτά, είναι, σαν κάτι, είναι κάτι σαν ευχολόγιο. Θα πρέπει να δούμε τι θα δοθεί από τον επόμενο προπολογισμό στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για να ελοπιθούν οι στόχοι. Ελπίζω ότι η στρατηγική αυτή δεν θα οδηγήσει σε επικράτηση των παλαιών κρατών μελών εντί των νέων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, θα σας συμβουλέψω κάτι. 15 επεξηγήσεις ψήφου είχαμε, ένα λεπτό η καθεμία αλλά έχουμε 53 συνολικά, 53 επεξηγήσει ψήφου. Άρα θα χρειαστεί πολλή χρόνο. Οποιοδήποτε θέλει να υποβάλει κάτι γραπτό είναι ευπρόσδεκτο. Με τα χαρά. Μία συμπληρωματική επεξήγηση ψήφου από τον κύριο Μπάλτσο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στατική για το 2020 και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ήταν κάτι που καταψήφισα εγώ διότι είναι προφανές ότι υιοθετεί μια νέα φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και εξηγεί και τονίζει ότι είναι κατά των προστατευτικών οικονομικών πολιτικών, δηλαδή κατά των κρατικών παρεμβάσεων. Αλλά θα έπρεπε να πάρουμε κάποια μαθήματα από τη χρηματοστική κρίση, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τις αγορές να κινούνται μόνες τους. Ε, είναι κάτι ορατό. Υπάρχει κάποιο, κάποια υπεριαλιστική προσέγγιση. Δηλαδή θα ισχύουν αυτομάτως οι κανονισμοί αν τα κράτη-μέλη ε, δεν φροντίζουν να θεσπίσουν την κατάλληλη νομοθεσία. Και θεσπίζεται και ευρωπαϊκή αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε άλλους τομείς φαίνεται με τέτοια προσέγγιση υποχρεωτικών νομικών δράσεων που θα δρομολογούνται και μειώνεται η αυτονομία των κρατών μελών. Γι' αυτό καταψήφισα. Η κυρία Γιάλα Σάντερ ε, πήγε σε κάτι και ήρθε εδώ να κάνει άλλη μια επεξήγηση ψήφου. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ε, ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να μιλήσω εκτός σειράς. Είχα κάτι επίγον στο γραφείο, έπρεπε να φύγω. Και ξέρετε, στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τα συζητήσαμε όσον αφορά τη ενόψη του 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο. Όμω, έχω μία επιφύλαξη που πρέπει να την εξηγήσω στου συναδέλφου. Στην παράγραφο 18, έτσι όπω έχει η διατύπωση, αφήνει κάποιες σκιές για κάτι που είναι αναλυθές. Δεν είναι σαφές ότι δηλαδή το Ελληνικό Συνέδριο επέκρινε κομισιόν και κράτη-μέλη για κάτι το οποίο καταρχήν ισχύει ως το αντίθετό του. Δηλαδή όχι για τη διαχείριση του 80% πρωτοβουλίου της Ένωσης, αλλά γιατί ακριβώς για πρώτη φορά φέτος μέσα σε μια δεκαετία μας έδωσε συγχαρητήρια το ελληνικό συνέδριο για το 33% και κάτι ε, που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και μιλούμε για τις αγροτικές δαπάνες και έγινε και ο έλεγχος καλύτερα τώρα. Οπότε, έτσι όπως διατυπώνεται, η διάταξη 18 προκαλεί σύγχυση σε όποιον το διαβάσει και λέει ότι επικριθήκαμε ενώ και το αντίθετο. Επομένως, θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί προς εσάς, συνάδελφοι, αλλά και προς τους Ευρωπαίους. Μανέσκο, είναι έκθεση Goldstone. Oh, I'm sorry, it's Nicole again. Ramona Nicole Manescu. Α, η κυρία, η κυρία Μανέσκου, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της έκθεσης Goldstone. Καταρχήν, φαίνονταν μια θετική πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό και ότι μας οδηγούσε στην πιο καλή λύση. Όμω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περισσότερο το Διεθνέ δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί διαπιστώνω ότι εδώ δεν χρησιμοποιεί τα διακριτήρια για Παλαιστίνους και για Ισραηλίτες. Αναφέρεται η Χαμάς ως μια τρομοκρατική οργάνωση και θεωρώ ότι όπως έχει αυτή η έκθεση δεν θα βοηθήσει στο να χαλαρώσει η ένταση στην ε, περιοχή. Άρα γι' αυτό και καταψήφισα. Πρόεδρος. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του δικαστή του κυρίου Γκόλστον είναι το έργο αξιοσέβαστων ανθρώπων που πρέπει να εμπιστευτούμε την κρίση τους. Δεν είναι πολιτική έκθεση και άρα πρέπει να εφαρμοστεί. Εγώ την υπερψήφισα, αλλά δεν συμφωνώ με όλα όσα αναφέρονται, παρά το ότι θεωρώ πως ήταν θετικό να υιοθετηθεί αυτή η έκθεση σήμερα στο Κοινοβούλιο και ελπίζω να συνεισφέρει ε, στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Η κυρία Ντρότς δεν είναι εδώ, οπότε περνάμε στην κυρία Κριστίνα Μπρουπάη. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δεκέμβριο του 2008 το Ισραήλ ξεκίνησε μια βάρβαρη επίθεση στην λωρίδα της Γάζας και ως αποτέλεσμα αυτού 1.400 άτομα πολίτες, ε, των οποίων 450 παιδιά πέθαναν. Η έκθεση Γκόλστον ε, ε, προσπαθεί να δει τα πράγματα αντικειμενικά και επεσήμανε αυτά τα εγκλήματα και επίσης έλεγε ποια στοιχεία του διεθνούς δικαίου παραβιάστηκαν από το Ισραήλ. Βεβαίως το κόμμα μας και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ της απόφασης του ΕΛΚ που αφορά την εφαρμογή των ε, συμπερασμάτων της έκθεσης και θα ήθελα να ζητήσω και συγγνώμη στα θύματα γιατί η κυβέρνηση του Ουγγαρία είναι κατά της έκθεσης ε, Γκολτσόν. Κύριε Φαντάλεν, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι μονομερής αυτή η έκθεση το γεγονός πως η Χαμάς ε, χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ως ασπίδα και τα σπίτια ως αποθήκες οπλισμού δεν το αναφέρει η έκθεση. Ίσως ε, αυτό οφείλεται γιατί η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ήταν υπό την Προεδρία της Σαουδικής Αραβίας, Λιβύης και το Πακιστάν, χώρες οι οποίες βεβαίως δεν είναι γνωστές για την ένδοξη δημοκρατία τους ή την ελευθερία γνώμης. Όποιος βεβαίως ανακατεύεται με αυτές τις χώρες, αυτά τα αποτελέσματα έχει. Δυστυχώς λοιπόν ψηφίσαμε κατά ολόκληρου αυτού του ψηφίσματος γιατί είναι πολύ μονομερής η έκθεση. Σας ευχαριστώ η κυρία Ρόιτεβα που σύρθηκε τα κουλά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε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 η πλειοψηφία στην Ολομέλεια εδέχθη την τοποθέτηση κατά του Χαμάς. Εξακολουθεί να απειλεί το Ισραήλ η Χαμάς. Γι' αυτό και το Ισραήλ πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του. Είναι λυπηρό το ότι θετήθηκε αυτή η μονομερής ημεροληπτική έκθεση. Και, και λυπάμαι που είχε τέτοια μεγάλη πλειοψηφία πίσω τη. Ελπίζω να μην επαναληφθεί στο μέλλον και η Ευρώπη να πολεμά για την ελευθερία τη έκφραση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επικρατεί τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ποιο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υποσχέθηκα να είμαι πιο σύντομο αυτή τη φορά. Νομίζω ότι ο δικαστής Γκόλστον δεν είναι ε, πραγματικά μερόληπτος. Καταψήφισα την έκθεση διότι θεωρώ ότι παρουσιάζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ε, μόνο σαν κάτι μαύρο και άσπρο, σαν μια σπρώμα Και η Ισραηλινή είναι κακή. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση κατά την άποψή μου. Πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιες μονομερείς μεροληπτικές κρίσεις. Εγώ, Πρόεδρε, και εσείς πήγαμε στην πόλη Σδέροντ που δεχόταν ε, τα πυρά ρουκετών της Χαμάς. Αυτή η έκθεση δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να περηφανεύεται στο μέλλον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω, δεν πήγα σε αυτή την πόλη, πήγα σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής, λέει ο πρόεδρο. Ο κ. Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά για την αναλογικότητα σε αυτή τη συζήτηση και διαρωτώ με οι αντίθετοι του Ισραήλ τι θεωρούν θα ήταν ανάλογη αντίδραση αν το εβραϊκό κράτος ε, τελικά βομβάρδισε με παρόμοιο τρόπο τη Γάζα κατά αναλογία των πυράβλων πέφτει στο Ισραήλ. Θα ήθελα να συζητήσω και την αναλογία, έλλειψη αναλογία στην έκθεση. Δημιουργείται το περίπου συνέστημα ότι διαβάζει κανεί τον κόσμο, να διαβάζει για μια βία επίθεση στην οποία ε, ξέχασε ότι γινόταν μια μάχη εκεί. Ε, ε, ήταν σαν να Ήταν απλώ μονομερή επίθεση. Δεν ξέρω ότι δεν πρέπει να επικρίνουμε το Ισραήλ. Έγιναν σφάλματα. Το Ισραήλ θέλει να βρεθούμε σε μια θέση όπου υπάρχει ένας καλός γείτονας, ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέλει αυτό και αυτή η πολιτική ε, μείωση των υποδομών καθυστέρησε το στόχο. Αλλά η μεροληψία και ο τόνο τη εκθέσεω, απ' την άλλη, απομάκρυνε περισσότερο την ιδέα τη λύση δύο κρατών. Ε, δηλαδή ένα Ισραηλινό κράτο και ένα Παλαιστινιακό κράτο που ζουν δίπλα-δίπλα σαν ε, ειρηνικοί γείτονε. Ευχαριστώ, κύριο Λάμσντορφ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το FDP σήμερα καταψήφισε το ψήφισμα πολλών ομάδων για την εφαρμογή της έκθεσης Goldstone. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια έκθεση στην οποία δεν υπήρχε καθαρή εντολή. Κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμφώνησε και επίσης εξισώνεται το Δημοκρατικό Ισραήλ με μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε διερεύνηση των συμβάντων. Κάθε άλλο. Πράγματι, το Ισραήλ πρέπει να ερευνήσει όλες τις ε, πτυχές ε, και εάν βρεθεί κάτι να δράσει ανάλογο. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει πως ε, πρέπει να εγκρίνουμε την πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ. Πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων και επίσης η επίσκεψη του Προέδρου Μπάιντεν δείχνει πως και η κυβέρνηση Ομπάμα παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη στην περιοχή και έχει την ε, στήριξή μας. Επίσης ακατανόητο είναι το ότι εγκρίθηκαν ακριβώς κατά την επίσκεψη αυτή νέοι οικισμοί από το Ισραήλ, κατά το οποίο βέβαια δικαίως πρέπει να επικρίνουμε. Ευχαριστώ. Περνάμε στην Λευκορωσία. Ο κύριος Νικολάτσιτς για ένα λεπτό. Ο κύριος Νικολάτσιτς λοιπόν, έχετε τον λόγο vážení Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δείχνει... δείχνει πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε αντίκτυπο στις ε, σχέσεις μας αν έχουμε καταπίεση και έλλειψη ε, κράτους δικαίου. Επίσης έχουμε και την υπόθεση με το ίντερνετ στη Λευκορωσία. Πρόκειται λοιπόν για καταπίεση, για έλλειψη ελευθερίας γνώμης, παραβίαση της δημοκρατίας και δικαιολογημένη είναι η δυσπιστία των πολιτών της Λευκορωσίας έναντι του κράτους τους πρόσφατα. Οι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης συνελήφθησαν και υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ της θέσεως ε, εν ισχύ των νέων μέτρων τον Ιούλιο που μας πέρασε και της θητείας του Επιτροπικών. Καληνός και για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτό το ψήφισμα, το προετοιμάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψηφίσαμε. Εμείς υπερψηφίσαμε το ψήφισμα εκφράσαμε την προθυμία μας να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα μειωνοτικά δικαιώματα στη Λευκορωσία είναι και μια απόδειξη ότι υποστηρίζουμε και την ελευθεροτυπία και την ελευθερία του λόγου που είναι θεμελιώδης αξία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χαίρομαι για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου που υποστηρίζει τη μειονότητα στη, την πολωνική μειονότητα στη Λευκορωσία, θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα για τους γείτονες και φίλους μας και να εξασφαλίσουν ότι τα μειονοτικά δικαιώματα γίνονται πλήρω σεβαστά στα κράτη-μέλη μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάσμαρε και έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι να ομιμοποιήσουμε την Ένωση των Πολωνών στη Λευκορωσία Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους τους πολίτες της Λευκορωσίας που δεν μπορούν να απολαύσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Έλαβα επιστολή ε, του πρεσβευτή της Λευκορωσίας στην Πολωνία χθε που ανησυχεί πολύ όσον αφορά τις προθέσεις των Ευρωβουλευτών που ήθελαν να υθετήσουν αυτό το ψήφισμα. Θεωρεί ότι δεν παρουσιάσαμε την κατάσταση αντικειμενικά στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, δεν αληθεύει αυτό. Πιστεύω ότι ε, το θέμα προχωρεί πιο πέρα. Μιλάμε εδώ για δικαιώματα των μειονοτήτων, ελάχιστα, ελάχιστες προδιαγραφές και είναι προς όφελος της Λευκορωσίας ε, που τα κάναμε όλα αυτά. Λαΐμα Λουτσία Αντρικίενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστήριξα το ψήφισμα όσον αφορά την κατάσταση κοινωνίας των πολιτών και εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία και σήμερα θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά τη σοβαρή μου ανησυχία όσον αφορά τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα προσφάτω στη Λευκορωσία κατά μελών τη κοινωνία των πολιτών, κατά μελών των εθνικών μειονοτήτων και των οργανώσεων αυτών. Και θα ήθελα να δηλώσω πλήρη αλληλεγγύη προς τους πολίτες που δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρως τα πολιτικά του δικαιώματα. Θα ήθελα να καταδικάσω και τη σύλληψη της Αγγέλικα Μπόρι, της Προέδρου της Ενώσεως Πολωνών στη Λευκορωσία και το Ανατόλιο Λεμπέτσκο που ήταν ηγέτης αντιπολίτευσης του, της, ε, του κόμματος των πολιτών και των Ηνωμένων Δημοκρατικών Δυνάμεων στη Λευκορωσία που είχε φιλοξενηθεί από το Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Και δυστυχώς για το λαό της Λευκορωσίας δεν μπορούν να αφεληθούν από πολλά προγράμματα και προτάσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα τμήμα της πολιτικής μας για την Ανατολική γειτονία. Πολιτική γειτονία. Ο κ. Στάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η κατάσταση στη Λευκορωσία μας υπενθυμίζει τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Αυτό το τονίζω γιατί μόλις είχαμε την πολύ λυπηρή ψηφοφορία για την έκθεση Goldstone. Οτιδήποτε σχετίζεται τον Κάφκασο, τη Λευκορωσία κτλ. Όταν τα συζητάμε αυτά τα θέματα πρέπει να θυμόμαστε την ελευθερία έκφρασης, ε, τη δημοκρατία. Αυτή είναι οι αξίες που έχουμε και πρέπει να τις προωθήσουμε και στη Λευκορωσία. Πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των θρησκευτικών μειονοτήτων που υφίστανται βιώσεις εκεί πέρα και να υπάρχει βεβαίως ε, ελευθερία άσκησης ε, της ε, θρησκείας. Ευχαριστώ. Αν Πρόεδρε, συμφωνώ με το μεγάλο μέρο του ψηφίσματο. Δεν ξέρω εάν δικαιούμεθα να λέμε στους Λευκορώσους τι πρέπει να κάνουν τη δημοκρατία τους και το δίθεν μα και εμείς εδώ είμαστε, είμαστε και εμείς ε, ε, δίθεν κοινοβούλιο κοιτάξτε είναι άδειο γύρω γύρω και τους λέμε ότι έχουν ενώθει εκλογέ και εμείς από την άλλη μεριά επίσης κάνουμε το ίδιο και παραπονιούμαστε επειδή εκεί πέρα οι απαράτσικ ζουν και βασιλεύουν ενώ εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τη, τη φοβερή μας αγροτική πολιτική και κορπορατισμό και συντεχνίες στην Ευρώπη. Ξέρετε τι έγινε. Όλοι αυτοί οι απαράτσικ και οι παλιοί κομμουνιστές ήταν αυτοί που ψήφισαν το ναι όταν τους καλέσαμε στην ε, Ευρωπαϊκή Σοβιετική Ένωση να μπουν και να προσχωρήσουν Θυμηθείτε το έργο του, του, του Orwell. Τι έγινε μετά με του ανθρώπου, τα ζώα και που τελικά δεν μπορούσε να, να καταλάβει ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι είναι ζώα στο έργο εκείνο του Orwell. Ο επόμενο. Πέραν του περιεχομένου, Πρόεδρε, εγώ, ε, ε, εγώ και επί της αρχή έχω αντίρρηση. Γάλλοι, Φλαμανδοί, Ούγγροι πατριώτε, Γερμανοί, Αυστριακοί διώκονται συνεχώ δικαστικά και πολιτικά και επαγγελματικά. Ενώ ε, το κοινοβούλιο εδώ πέρα αδιαφορεί ή συμπλέει με τους διώκτες διακόπτη ο πρόεδρος εγώ σας ακούω στα φιλανδικά από το κανάλι της Διερμίας Αγγλικής το οποίο δεν είναι τόσο ε, δόκιμο <laughs> οπότε αν μπορείτε διορθώστε Merci. Est-ce que ça va comme ça, Monsieur le Τώρα με ακούτε, Πρόεδρε. Πρόεδρε, σας έλεγα ότι οι πατριώτες σε Γαλλία, Φλάνδρα, Ουγγαρία, Αυστρία διώκονται δικαστικά, επαγγελματικά, πολιτικά. Με την αδιαφορία και το πράσινο φως που είναι στο κοινοβούλιο στο και αυτό γίνεται πάντως σε όλο τον κόσμο και εκτός των συνόρων μας. Να και χθες είχαμε και εκείνη την, ε, το ψήφισμα για την Ουγγαρία για την Ουκρανία και πάρα πολλοί πατριώτες ε, Ουκρανοί Θεωρούν ότι ο Στέπαν Μπαντέρα που είναι εθνικός ήρωας προσβάλλεται. Γιατί τι να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ του, του, των δύο ολοκληρωτισμών της Εκκλησίας και του Σοβιετικού ολοκληρωτισμού. Και εμείς τους ταπεινώνουμε. Νίκ Γκρίφιν είναι πραγματικός πατριώτης είναι ό,τι και για μας η Ιωάννα της Λορένης. Άρα θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να σέβεται τους ήρωες και των άλλων ξένων χωρών. Right. that section. We've got about halfway through. Λοιπόν, τα μισά κάναμε περίπου, έχουμε άλλο ένα μισάωρο περίπου. Πάμε στη φορολόγηση και οικονομικές συναλλαγές. Πρώτος ομιλητής στο ECR για δύο λεπτά είναι η κυρία Σβίνμπεργκ, Ευχαριστώ. Το ECR αναγνωρίζει ότι οι χρηματοστατικέ υπηρεσίε και ο τομέα αυτό των χρηματοστατικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αναμένει να ξεφύγει αλόβητο από την κρίση λόγω τη προσοχή έγιναν πολλέ ζημιέ και τι ζημιέ πρέπει να τι πληρώσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Τα νέα συστήματα θα πρέπει να δημιουργηθούν να εξασφαλίσουμε ότι θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και οι πόροι θα διατίθενται για κατεπίγουσε ανάγκε, για να σταθεροποιούνται συστημικά προβλήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο ότι στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών ότι ήρθε η ώρα τώρα για, κάποιες, ε, για κάποιο φόρο των οικονομικών συναλλαγών. Όποιε αμφιβολίε και αν υπάρχουν για την πρακτικότητα αυτού του μέτρου, και αυτού του συστήματο κανένα μέτρο δεν πρέπει να αποκρίνεται από τη στιγμή που θα έχει την υποστήριξη όλη τη διεθνού κοινότητα και από τη στιγμή που έχουν ρήτε διαφύλαξη, ούτω ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να μην μπορεί να αποφευθεί το σύστημα. Τα περισσότερα ψηφίσματα σήμερα τα υποστηρίξαμε. Εξαιρείται όμω παράγραφο 7 του, του ψηφίσματο που υποστηρίζουμε. Είμαστε αντίθετοι όσον αφορά το να έχει εξουσίε προσθέτων φόρων η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτή η παράγραφο διατείνεται ότι αυτό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και δεύτερον, το όλο θέμα των οικονομι... του φόρου οικονομικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να συλλέγονται για αγαπημένα προγράμματα χρήματα, όσο αξιόλογα και αν είναι. Θα πρέπει ανταυτού να εξασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα και να προστατευτούμε έναντι γεγονότων που οδήγησαν στο πρόσφατο οικονομικό χάος. Αυτό το ψήφισμα ω έχει εστιάζεται πολύ στη λύση του φόρου συναλλαγών και ότι θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συλλέγει του φόρου και τα κράτη-μέλη και τα χρήματα να χρησιμοποιούνται για προγράμματα για καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο και αντί να σταθεροποιείται ο οικονομικό τομέα και προτείνει ότι αυτό ο φόρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μπορεί να είναι εφικτό χωρί γενική ε, συμμετοχή. Γι' αυτό καταψηφίσαμε το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ευχαριστώ. έχει το Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, απήχα εγώ στο ψήφισμα για τις δημοσιονομικές συναλλαγές γιατί δεν αρκεί για να καταπολεμήσει την χιδαία αντικοινωνική κερδοσκοπία από τις λεγόμενες ε, σεβαστές τράπεζες όπως η Goldman Sachs. Υπήρχε στις 8 Φεβρουαρίου ένα δείπνο στη Νέα Υόρκη από επικεφαλής 8 hedge funds που σκόπευαν να επιτεθούν στο ευρώ και οι καρχαρίες αυτοί που ελέγχουν άνω των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ σχηματίζουν κατά του ευρώ και της Ελλάδας ιδιαίτερα για να κερδίσουν οι ίδιοι. Και μάλιστα η Κομισιόν όχι μόνο δεν σηκώνει ένα δάκτυλο για να του σταματήσει, αλλά τι κάνει. Συνεννοείται μαζί τους και πιέζει τους καημένους στοχούς εργαζόμενους στην Ελλάδα για να ωφεληθούν αυτά τα παράσιτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει δημόσια διευθυνσία και δημοκρατικός έλεγχος των hedge funds και των επενδυτικών τράπεζων για να γίνουν έργα, για να ωφεληθεί η κοινωνία και να μην καταστρέφει η κοινωνία για χάρη του, της απληστίας. Ο κύριος Μποργέζιο, έχουμε αλλά ήθελα να, ήθελα να είμαι κατά τη πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστεί ένα φόρο, να θεσπιστεί ένα φόρο. Όπω δείχνουν οι δηλώσει του κυρίου Σεμέτα, οι πρόσφατε δηλώσει στο European Voice, ότι θέλει να επιβάλλει ελάχιστο το ε, φόρο όσον αφορά αυτέ τι συναλλαγέ. Εμεί δεν θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε δυνατότητα να επιβάλλει άμεσου φόρου. Είναι ένα προνόμιο μη συνταγματικό που ανήκει στα κάτι μέλη κανονικά παραβιάζει το no taxation without representation, αυτή την αρχή. Εμεί θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια να εισαχθεί μια άμεση φορολόγηση. Και έχουμε και την απόφαση του 2009 του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας πάνω σε αυτό. Ήδη είδαμε μια πρώτη γεύση από τον Βον Ρομπουί, όταν σε μια μυστηριώδη συνεδρίαση που έγινε μια εβδομάδα πριν από το διορισμό του στην ομάδα Bildenberg που δεν λειτουργεί με μεγάλη διαφάνεια αυτή η ομάδα, ανακοίνωσε ότι λαμβάνω την υποχρέωση να προτείνω άμεσο ευρωπαϊκό φόρο όσον αφορά τον άνθρακα, του δεξιού του άνθρακο, που θα αύξηνε τα, την τιμή των καυσίμων των υπηρεσιών, άρα ει βάρο των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η πρόταση του ευρωπαϊκού φόρου φορολόγηση είναι κάτι μη συνταγματικό, αντί συνταγματικό. Ευχαριστώ. Ο κ. Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πιστεί ότι χρειάζεται ένας φόρος για τις οικονομικές συναλλαγές. Δέχομαι όμως τα ειλικρινή κίνητρα εκείνων που υποστηρίζουν την πρόταση. Είναι ένα θέμα όπου ίσως να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εκείνων που έχουν ειλικρινή διάθεση, ειλικρινές προθέσεις. Όμως δεν μπορεί να επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος επουδενή αποκλειστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας φόρος Τόμπιν που θα εφαρμοζόταν μόνο περιφερειακά θα οδηγούσε σε μια φυγή κεφαλαίων που θα πηγαίνετε κεφάλαια εκεί που δεν υπάρχει φόρος. Γιατί υπερψηφίστηκε με τέτοια διαφορά ένα τέτοιο σύστημα που θα φέρει σε δυσμενή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Επετίθεται κατά των τραπεζών, κατά του Λονδίνου, του Σίτι και έχει ανεξάρτητη πηγή εσόδων Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να προσφύγει στα κράτη-μέλη. Τα δει κανεί όλα αυτά μαζί, μαζί με τι άλλε προτάσει που έρχονται για εναρμόνιση τη οικονομική εποπτεία, η οδηγία για αναλεκτική διαχείριση των πόρων, βλέπουμε ότι απειλείται το City του Λονδίνου και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θα καταλήξει στην παινία. Ευχαριστώ και ο Σκαμάλ έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όποιος κοιτάξει την πρόσφατη κρίση θα αναρωτηθεί πώς ε, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση όπου λέγαμε ότι οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν και δισεκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων στήριζαν αυτές τις τράπεζες. Οπότε όταν σκεφτόμαστε αυτή την ιδέα του παγκόσμιου φόρου Φαίνεται λογική αν είναι να βοηθήσουμε τα θύματα των κρίσεων αλλά και αυτούς τους φτωχότερες χώρες. Αλλά εάν δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό και το, τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχει, εάν δούμε τι θα γίνει όντως στις αγορές, τι θα συμβεί. Οι τράπεζες θα περάσουν το κόστος στους πελάτες τους. Επίσης θα επηρεάσει ε, όσους θέλουν να εμπορευθούν με τις αναψώμενες χώρες και τις αναψώμενες χώρες στο εμπόριό τους με τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια υπάρχει και το κόστος της ασφάλισης που είναι πολύ μεγάλο στο διεθνές εμπόριο. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να δώσουμε δισεκατομμύρια από τους φόρους μας σε διεφθαρμένες ε, κυβερνήσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρηματίες στις φτωχές χώρες για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ενιαία Ευρωπαϊ... στον νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών, κ. Πασκά. Ďakujem za slovo, pán vážený pán predsedajúci. Chcem oceniť eh, úsilie Európskej únie o zavádzanie... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ενίο καθιστός τραπεζικής πληρωμές στην ε, Ευρώπη. Από την άλλη βλέπουμε πως υπάρχει κατάχρηση από τις τράπεζες ε, του κανονισμού αυτού και βεβαίως ε, τα τέλη προσαρμόστηκαν όσον αφορά τις πληρωμές έτσι ώστε να είναι ίδια με το κόστος του εσωτερικού αλλά ταυτόχρονα επιβάλλονται νέα τέλη για μεμονωμένες εναλλαγές στα υποκαταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό με την εισαγωγή του νέου κανονισμού δεν καταργήθηκαν αυτά τα τελευταία τέλη, οπότε εξακολουθούν να κάνουν κατάχρηση της κατάστασης οι τράπεζες. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε σε ποιο βαθμό ο νέος κανονισμός θα τηρηθεί από τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Περνάμε στην καταπολέμηση της πειρατείας. Ο κ. Κραμός για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ψήφισα για την έκθεση και την καταψήφισα γιατί δεν θέλω κάτι να ψηφίζεται και να εγκρίνεται πίσω από τις πλάτες των ε, εκλογέων, των ψηφοφόρων μας. Έχει αυξημένε αρμοδιότητε με τη συνήθεια στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να φροντίσει να είναι σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε εγκρυπτό και απαραβίστο τέτοιε συμφωνίες. Αυτό αντιβαίνει στο κοινωτικό δίκαιο. Και δυσκολεύει. Τι, το, το, να ξεκιώνονται με το κοινωτικό δίκαιο οι Ευρωπαίοι. Οπότε με μεγάλη μου χαρά βλέπω να έχει τέτοια απόκριση και ανταπόκριση το Κοινοβούλιο στις προτάσεις κομισιών για αυτά τα παραπημένα προϊόντα και τις απομιμήσεις. Η επομένη κυρία. Σε σχέση με αυτές τις απομίσεις εμπορικών προϊόντων, νομίζω ότι έγιναν κρυπτό χωρίς καμία διαφάνεια αυτές οι συμφωνίες, κάτι το οποίο αντιβαίνει στη, στην παράδοση τη δημοκρατική, την παράδοση της ε, διαφάνειας που προσδοκούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει έλεγχος και είναι για κάτι το οποίο αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πάντως, όσον αφορά το περιεχόμενο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον επόπτη για τα δεδομένα, γιατί ε, έχει διατυπωθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχει διάλογο για το άκτα με διαφάνεια. Δεν είναι δυνατόν πάντως τα εμπορικά συμφέροντα να κατησχύουν των ατομικών δικαιωμάτων ή της ελευθερίας έκφρασης ή του δικαιώματος στο δικαστή. Προσοχή να μην νομοθετούμε με τρόπο που περιορίζουμε τις ελευθερίες, τι ατομικέ και τα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει και, το, και η Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο να φροντίσουν να υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο και διαφάνεια. Ο κ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάτι σημαντικό που υπάρχει για το ψήφισμα, για την πρόταση ψηφίσματο ήταν το γεγονό ότι καταφέραμε να πετύχουμε συμμαχία στο Κοινοβούλιο και ήταν ένα τομέας κοινή συμφωνία, δηλαδή εν πληροφοριών σωστών που αφορούν τι διαπραγματεύσει. αυτό που έβλεπε κανεί στα μπλοκ ήταν εφήμε και προτάσει όπω η κατάσχεση φορητών υπολογιστών ή μηχανημάτων ε, που παίζουν MP3 στα σύνορα. Εμεί θέλαμε πληροφορίε, θέλαμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη συμφωνία αυτή ε, αντιπαραποίηση, αντιπειρατεία. Ο επίτροπο εχθέ πήρε το μήνυμα, ήταν ηχηρό και χαίρομαι που υποσχέθηκε να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται εκ μέρου 27 κρατών μελών και εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ενώσεω, είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η διαπραγματευτική θέση και θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση αντικτύπων ε, για τα προτινόμενα. Πώ θα επηρεαστεί η βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Καλωσορίζω τα σχόλια του Επιτρόπου που ακούστηκαν στο βράδυ και προσβλέπω σε περισσότερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πάσκα για ένα λεπτό. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενισχώ πάρα πολύ για τη συμπεριφορά της Κομισιόν όσον αφορά αυτή τη συμφωνία διαπραγματεύσεις γίνονται ε, και κλεισμένων των θυρών. Οι ευρωβουλευτές δεν ε, έχουν πληροφόρηση. Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αναμένει η Κομισιόν να φέρει μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευθύνη. Δεν είναι μήνυμα αυτό για την κοινή γνώμη, ούτε και για τον υπόλοιπο κόσμο εάν θα πρέπει να επεξεργαστεί μετά πολλέ φορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση την συμφωνία. Δείχνει πώ δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Thank you. Next we come to... Ε, ευχαριστώ. Ε, Γενικευμένε Ο κ. Καμάλ έχει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, το σύστημα που έχουμε το GSP πρέπει να αναθεωρηθεί των δασμολογικών προτιμήσεων και το παρόν σύστημα εκπνέει. Και ένα από τα πράγματα που είναι σημαντικά όταν εξετάζουμε αυτό το σύστημα και το CSP Plus είναι ότι κατά τη των πραγματεύσεων επί των συμφωνιών οικονομική συνεργασία και εταιρικών σχέσεων, πολλά κράτη-μέλη σε διάφορε περιφέρειε ήταν κατά υπογραφή συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι που επέκρινα όσον αφορά αυτέ τι συμφωνίε εταιρική είναι ότι χρησιμοποιούσαν την κοινή προσέγγιση για όλου. Και αυτό που με ανησυχήσε ήταν κατά τη διάρκεια συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάλληλο είπε ότι οι οικονομικέ αυτέ συμφωνίε εταιρική σχέση δεν είναι μόνο για εμπόριο, αλλά για εξαγωγή του προτύπου τη περιφερειακή ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Υπάρχουν διάφορε χώρε που θέλουν να έχουν συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να μπορούν να εξάγουν αγαθά και υπηρεσίε του σε εμά επί προτιμησιακή βάσεω. Γι' αυτό αυτό που θα πρέπει να προταθεί θα είναι να προσφέρουμε σε αυτέ τι χώρε που θέλουν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία αλλά δεν ταιριάζουν τα κριτήρια τη εταιρική τη σχέση να προσφέρουμε το GSP Plus συν σαν μια εναλλακτική λύση. Να είμαστε πιο ευέλικτοι. Έτσι οι επιχειρηματίε θα δημιουργήσουν πλούτο και θα βγάλουν του στοχού από τη φτώχεια σε πολλέ από αυτέ τι χώρε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χάναν. And... Η Νότια Αμερική και η Λατινική Αμερική μπαίνουν σε μια ε, σε ένα κράτος που επικρατεί. Βλέπουμε ότι είναι καθεστώτα αυταρχικά. Δεν είναι ακριβώ δικτατορικά καθεστώτα, αλλά δεν υποστηρίζουν την κοινοβουστική δημοκρατία. Δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Και αυτοί που εκλέγονται τελικά διαλύουν διάφορες, ε, το ανώτατο δικαστήριο, τα, τις βουλές, ε, διαλύουν ε, τα συντάγματα και ετοιμάζουν καινούρια συντάγματα. Και ακολουθούν σοσιαλιστικές αρχές. Και ποιο επιλέγει να, επι, να επικρίνει αριστερά και ένα από τα λίγα καθεστώτα που απολαμβάνει λαϊκή υποστήριξη του Αλβάρου Ρίρε στην Κολομβία που έχει την υποστήριξη πάνω από τρία τέταρτα του πληθυσμού διότι κατέστησε την τάξη σε αυτή την άτυχη χώρα και επευλήθη στις παραστατικές οργανώσεις της αριστεράς και της δεξιάς. Δείχνει ότι έχει εξαιρετικές προτεραιότητες. Εκείνος θα έπρεπε να είναι και είναι περίεργο που διάλεξαν προτεραιότητα να του επιτεθούν οι περισσότεροι εδώ. Είναι ντροπή το, το να κοφεύουμε και να παίζουμε το παιχνίδι φυσικά των παραστρατιωτικών. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Αλμπερτίνη για την έξοχη δουλειά που έκανε επ' αυτού του θέματος που είναι πολύ σημαντικό την Ευρωπαϊκή Μετά στη ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα. οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και κοινή ασφάλεια αυξήθηκαν και πιστεύω ότι εδώ πολλοί θέλουμε μεγαλύτερες ευθύνες και μεγαλύτερη συμμετοχή όσον αφορά την εξωτερική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμμερίζομαι την πρόσκληση που απευθύνεται προς την ύπατη εκπρόσωπο για την ΚΕΠΑ να διαβουλευτεί με την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ευκαιρία του διορισμού για τις θέσεις των διαφόρων μελών της εξωτερικής υπηρεσίας για εξωτερική δράση και την επέκταση της πρόσβασης στις πληροφορίες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τις πληροφορίες πέρα από το Συμβούλιο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα πρόοδο αυτά που αναφέρονται εδώ για μια πολιτική εξωτερική τη Ευρωπαϊκή Ενώση που θα είναι ισχυρή και να παίξει το ρόλο τη στο σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβάλλει το βάρο τη στο διεθνέ προσκήνιο. Ευχαριστώ. Σίνκλερ, επόμενο αγορητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καταψήφισα τις τροπολογίες 17 Δέλτα και 17 Δέλτα και 19 που κατηγορούσαν τον ΝΑΤΟ και έλεγαν να φύγουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα τελευταία επιχειρήματα όσο πιστεύουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι πως η Ευρώπη τι κράτησε την ειρήνη εδώ πέρα στην Ευρώπη τα τελευταία 60 χρόνια. Όχι. Το ΝΑΤΟ διατήρησε την ειρήνη. Και είναι ντροπή να υπερψηφίζονται τέτοιες τροπολογίες. Βλέπω πως αυτοί που, ψώ, που πρότειναν, με την τροπολογία είναι απομεινάρια μιας αποτυχημένης ιδεολογία που κρατούσαν τους ανθρώπους πίσω από τύχη. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ προστάτευαν την Ευρώπη από αυτό τον εφιάλτη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να γραφτεί στα πρακτικά της ΕΠΑ, τον Καναδά, και τις λοιπές χώρες μας προστάτευσαν, προστάτευσαν η ελευθερία μας και είναι προς το συμφέρον μας να ενωθούμε αυτές τις χώρες κατά της νέας απολυταρχίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στην αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Ο κ. Αντωνιώτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα διότι ήθελα να υπογραμμίσω ότι θέλουμε αύξηση των συνεργειών και της συνεργασίας στο στρατιωτικό και πολιτικό τομέα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών. Θα πρέπει να σεβαστούμε όμως και κάποιες ουδέτερες θέσεις. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτηση. Γενικά είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί συντονισμού με ένα κέντρο επιχειρησιακό μόνιμο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω υπό την αιγίδα τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου για την ΚΕΠΑ που θα επιτρέπει αποτελεσματικό συντονισμό του κοινού σχεδιασμού των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων και για να εξαλειφθούν προβλήματα της λειτουργίας και καθυστερήσεις που δυστυχώς ε, αντιμετώπισε το τρέχον σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Καταψήφισα τη σχετική έκθεση γιατί επαναλαμβάνει τις επικίνδυνες κατευθύνσεις που έδινε η, η συνθήκη της Λισαβόνας για την ευρωπαϊκή στρατηγική της άμυνας και της ασφάλειας. Απαιτεί δηλαδή τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επεμβάσεις, αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ και τη στενή σχέση μαζί του και ακόμα οθεί και μάλιστα σε συνθήκε κρίση και μεγάλων κοινωνικών αναγκών στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. κατά την άποψή μου η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή δηλαδή τώρα που κρίνεται η αρχιτεκτονική του κόσμου να ακολουθήσει φιλιρινική πολιτική και μια άλλη πολιτική αντίληψη για την ασφάλεια να ακολουθήσει ανεξάρτητη και χειραφετημένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική από τι ηνωμένε πολιτείε να επιδιώκει τη διευθέτηση των διεθνών διαφορών με πολιτικά μέσα και να πρωτοστατεί στο σεβασμό του διεθνού δικαίου και του ενισχυμένου ρόλου του οηε. αυτή η πολιτική νομίζω ότι εκφράζει καλύτερα του ευρωπαίου πολίτε. σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Διακόπτη συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τους διερμηνείς.